κύριοι, οι αρμόδιες Ιταλικές αρχές ε, μου γνωστοποίησαν ότι ο κύριος Ροζάριο Κροτσέτα από την 17η Δεκεμβρίου 2012 διορίστηκε ως πρόεδρος της περιοχής της Σικελίας και από την κυρία Φραντσέσκα Μπαρατσού αντικαθίσταται. Εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας για την εκλογή του στον συνάδελφο ε, Κροτσέτα και για την ε, ε, εισαγωγή ενό ε, βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σύμφωνα με το άρθρο του κανονισμού από τη 17η Δεκεμβρίου διαπιστώνεται η χειρία της ε, έδρας του και διαπιστώνουμε ότι η κυρία Φραντσέσκα Μπαρατσού εισέρχεται ως μέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλωσορίζουμε την κυρία Μπαρατσού και σύμφωνα με το άρθρο 3, εδάφιο 2 του κανονισμού θα συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα στι συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου και των οργάνων του εφόσον δεν θα έχει δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση σε αφορά την εντολή της και υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι θα έχει δηλώσει ότι δεν έχει κάποιο αξίωμα το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με την εξαγωγή των καθηκόντων της ως Ευρωβουλευτού σύμφωνα με τον κανονισμό. Η κυρία Φρίντα Μπρέπολς μας ανακοίνωσε την υπαναχώρησή της, την αποχώρησή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την 31η Ιανουαρίου 2013. Λαμβάνουμε υπόψη αυτή τη δήλωση και σύμφωνα με το άρθρο 4 εδάφιο 3 θα υπάρξει χειρία της έδρας από αυτή την ημερομηνία. Οι αρμόδιες βουλγαρικές αρχές μας ειδοποίησαν για την εκλογή του κυρίου Πρέσλαφ Μπόρισοφ από την 1η Ιανουαρίου 2013. Ο κύριος Μπόρισοφ θα αντικαταστήσει την κυρία Ηλιάνα Ιβάνοβα. Καλωσορίζουμε τον νέο συνάδελφο και υπενθυμίζουμε ότι ο κύριο Μπορισόφ, σύμφωνα με το άρθρο 3, εδάφιο 2 του κανονισμού, με πλήρη δικαιώματα θα συμμετέχει στι συνεδριάσει του Κοινοβουλίου και των οργάνων του, εφόσον ε, δεν θα έχει υπάρξει ε, κάποια ένσταση σε σχέση με την εντολή του. Και θα έχει δηλώσει προηγουμένως ότι δεν θα έχει κάποιο αξίωμα το οποίο να έρχεται σε σύγκρουση με την άσκηση των καθηκόντων του ως Ευρωβουλευτού δεν θα έχει κάποιο αξίωμα το οποίο θα είναι ασύμβατο με την ιδιότητά του αυτή. Οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές γνωστοποίησαν ότι ο κύριος Τζόρτζε Μπεκάλι ή Μπέκαλη, δεν ξέρω πώς προφέρεται, από την 19 Δεκεμβρίου 2012 εξελέγει στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού διαπιστώνει την χειρία της έδρας του ε, συναδέρφου και θα ειδοποιηθεί η αρμόδια αρχή και για την εκλογή, από ε, την εκλογή του κυρίου Ντουμίτρου Σαμφιρέσκου μας ε, ειδοποίησαν οι ρουμανικές αρχές. Ο κύριος Σαμφιρέσκου θα αντικαταστήσει τον κύριο Μπεκαλή και καλωσορίζουμε τον νέο συνάδελφο και υπενθυμίζουμε και πάλι εδώ ότι για τον κύριο Σαμ Φιρέσκου θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες και διατάξεις του κανονισμού. Θα συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα στις συνεδριάσεις του Ευρωκοινοβουλίου και των οργάνων του υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει δηλώσει ότι δεν έχει κάποιο αξίωμα το οποίο να συγκρούεται με την ιδιότητά του ως Ευρωβουλευτού και που δεν θα είναι ασύμβατο με αυτή την ιδιότητά του. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έθεσαν αίτημα για την άρση τη ασυλία του Ευρωβουλευτού κ. Σπύρου Δανέλη. Σύμφωνα με το άρθρο 6, εδάφιο 2 του κανονισμού, αυτή, αυτό το αίτημα θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Η Νομική Επιτροπή, στη συνεδρίασή τη στι 17 Δεκεμβρίου 2012, εξέτασε την ε, εντολή νέων μελών και ομόφωνα